Η Ιταλία φυσικά έσωσε την Ευρώπη στο παρελθόν και την τιμή της Ευρώπης. Αλλά δεν λύνουμε έτσι το ζήτημα υπερασπιζόμενη την τιμή της Ευρώπης. Γιατί όποιο κράτος βρεθεί στη δινή θέση της Ιταλίας φτάνει σε ένα σημείο κορεσμού. Οι μηχανισμοί ένταξης δεν λειτουργούν πλέον. Οι επαναπατρισμοί είναι δύσκολοι γιατί δεν είναι αποδοτικοί. Δυστυχώς με ορισμένες χώρες δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τους μετανάστες. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο διμερός πολλές φορές. Άρα αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει ούτε επαναπατρισμός. Γι' αυτό αυτό φτάσαμε σε μια πιο αυστηρή στάση. Το λέμε. Το λέμε ανοιχτά. Με σαφήνεια και διαφάνεια. Γιατί θεωρήσαμε, αφού καταρτήσαμε αυτή τη διαρθρωμένη στρατηγική, ότι δεν μπορεί να γίνει πάγια τακτική. Δεν είναι ο μόνος δρόμος αλλά ένας δρόμος για να σταματήσουμε την διακίνηση ανθρώπων. Υπάρχει μεγάλη υποκρισία στην Ευρώπη. Οι μετανάστες γίνονται πρόβλημα όταν τους βλέπουμε με τους προβολείς στη Μεσόγειο, όταν Μίκιο το κάνει θέμα στα ΜΜΕ. Αλλά μην ξεχνάμε τους μετανάστες εκεί όπου άφησαν το χωριό τους και όπου τους αναλαμβάνουν οι διακινητές. Ξέρετε πόσο στοιχίζει αυτή η, πορεία της ελπίδας μετά από βασανισμούς, μετά από μεγάλα βασανιστήρια, 3.500 δολάρια το ελάχιστο. Μιλάμε για φτωχούς ανθρώπους που έχουν μεγάλη δυσκολία να βρουν αυτά τα χρήματα και στη συνέχεια τους αποσπώνται και αντιμετωπίσουν μύρια όσα δεινά. Η Ιταλία μέσα στα πλαίσια του Search and Rescue σε αυτή τη διαδικασία διάσωσης προσπάθησε πάντα να τηρήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ισχύει και στην περίπτωση Διτσότη, γιατί είδαμε τους πιο ευάλωτους, τους ε, πήραμε και τους μεταφέραμε στη γη. Όπως και στην τελευταία περίπτωση, είχαμε ένα πλοίο όπου ζητήθηκε η υγειονομική περίθαλψη, είδη διατροφής και μετά από ημέρες στο λιμάνι προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κακή μεταχείριση, αλλά φτάσαμε σε κοινά συμπεράσματα σε επίπεδο 28 και δεν μπορείτε ε, να λέτε ότι υπάρχει μηχανισμός επανακατανομής. Δεν λειτουργεί έμπρακτα αυτός ο μηχανισμός. Δεν είναι υποχρεωτικός για όλους ας φτάσουμε και σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Υπάρχει ασφαλές λιμάνι μόνο όταν αποβιβάζεται κανείς στην Ιταλία, μα δεν είναι το πιο κοντινό λιμάνι, το πιο σίγουρο. Ο μηχανισμός επανακατανομής δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο σε τρεις, τέσσερις, πέντε χώρες πρέπει να συμμετέχουν όλοι σε αυτό το μηχανισμό αλληλεγγύης. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα. Μην το κρύβουμε. Υπάρχουν χώρες που λένε ότι είναι ε, διαθέσιμες να συμμετάσχουν στο μηχανισμό επανακατανομής, αλλά το κάνουν μόνο για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασίες. Κανένας δεν θέλει τους οικονομικούς μετανάστες. Παραμένουν στα λιμάνια αποβίβασης. Τώρα, για την οικονομία και για τις επενδύσεις και τις υποδομές, είπατε ότι η Ιταλία δεν θέλει να κάνει τις σωστές μεταρρυθμίσεις. Καλύτερα να πληροφορηθείτε γι' αυτό, γιατί στη διαδικασία διαμεσολάβησης με τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον αντιπρόεδρο, τους αντιπροέδρους Ντομπρόφσκης και Μοσκοβισή από την πρώτη φορά που τους συνάντησα. Δεν τους είπα να μην μπούμε στη διαδικασία επί παραβάση. Τους έδωσα ένα κόρπους όπου αναφέρονται όλες οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει. Και είπαμε ότι η Ιταλία, και είπαμε ότι δεν ισχύει ότι η Ιταλία δεν θέλει να κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε εγκρίνει και υλοποιούμε ένα ογκοδέστατο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ε, περισσότερο από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Παρακαλώ, κατά την ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα κάνετε τι ερωτήσεις σα. Εγκρίναμε νόμο κατά της διαφθοράς που προβλέπει πρότυπα ε, κατά τη διαφθορά από τα πιο απαιτητικά, όχι μόνο στην Ευρώπη, Κύριε Ντάντε, αν θέλετε να μιλήσετε μετά, μετά. Μην διακόπτετε τώρα παρακαλώ φωνάζοντα. Παρακαλώ. Δεν μπορεί να γίνεται διάλογο μονομερής. Με το χρόνο που χάνουμε με τι διακοπέ, δεν θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτέ. Προσπαθώ να απαντήσω. Θα απαντήσετε μετά, θα απαντηθούν μετά οι ερωτήσει. Με τα απαιτητικότερα λοιπόν πρότυπα κατά τη διαφθορά, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά διεθνώ, έχουμε προβλέψει μια μεταρρύθμιση ρίζοσπαστική για την περίπτωση τη πτώχευση. Στην ε, Ιταλία δεν ε, γίνεται πια λόγο για πτώχευση ε, γίνεται λόγος για κώδικα των εταιριών που χρειάζονται διάσωση. Μιλάμε για ένα ογκοδέστατο σώμα άρθρων. Θα πρέπει εδώ να δούμε τα σχετικά διατάγματα που χρειάζονται, τα νομοθετικά διατάγματα, για να απλοποιήσουμε όλες τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά. Πρέπει να γίνουν πιο ε, ταχείες οι όλες διαδικασίες. Αυτό έχουμε αρχίσει να το επιδιώκουμε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε καταξιοδότηση πράξη και θα κοιτάξουμε να γίνει ροζοσπαστική ε, μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για τους δημόσιους διαγωνισμούς, τις προμήθειες. Έχουμε και άλλον νόμο για τον αστικό κώδικα, για την ε, εκδίκαση των υποθέσεων στα ποινικά δικαστήρια. Αυτά κάνουμε. Όταν λέτε ότι είμαστε κατά των επενδύσεων, μα τι να πω, παρακολουθείτε άλλες συζητήσεις, ακούτε να μιλάνε άλλοι. Ε, με συγχωρείτε, αλλά το πρόγραμμα για τις επενδύσεις στις υποδομές στην Ιταλία. Το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει τις τα τεράστια κονδύλια που προβλέπονται για τις επενδύσεις, τα 13 δις πέραν των κρατικών επιχειρήσεων οι οποίε, όπω λέτε ε, έχουν έρθει παρόλα αυτά να συζητήσουν μαζί μα στο Μεγαροκίτσι. Εδώ λοιπόν κοιτάζουμε ένα πρόγραμμα ασφάλεια για όλη τη χώρα. Ένα εθνικό πρόγραμμα για, τις, ε, για τους κινδύνους υδρολογικού χαρακτήρα. Κοιτάζουμε να προστατεύσουμε τι υδάτινες, τι υποδομές μας για την υδροδότηση. Και εδώ χρειαζόμαστε και ευελιξία. Το, συναντηθήκαμε το συνεννοηθήκαμε με την Επιτροπή και το αποσπάσαμε. Τρία δις. Τρία δις 200 εκατομμύρια επιπλέον πέραν του επενδυτικού προγράμματος που ήδη έχει οριστεί, χρειαζόμαστε. Πρέπει να ακούσουμε και τις διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να υπάρχει διαφορά απόψεων. Στη δημοκρατία αυτό είναι το ωραίο, ότι υπάρχουν συζητήσεις για τα κοινά δημοσίω, οπότε ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Όμως το να αγνοεί κανεί όλα αυτά σημαίνει ότι ουσιαστικά ε, κοροϊδεύει τους ε, Ευρωπαίους πολίτες, όχι μόνο τους Ιταλούς. Σε ό,τι αφορά την ΤΑΒ, Τότε αφορά λοιπόν τα γρήγορα τρένα, είναι ένα πρόγραμμα που ήδη εγκρίθηκε. Ε, η κυβέρνηση ήδη θεωρεί ότι είναι ορθό απέναντι στις ανάγκες των πολιτών, ακριβώς επειδή επιπλέον υπάρχουν και αξιολογήσεις ε, που δικαιολογούν αυτό το έργο. Εδώ και 25 χρόνια υπάρχουν. Τώρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να υλοποιηθεί. Ε, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η προκαταρκτική φάση, αλλά πριν αρχίσουμε να εκτελούμε και να χρησιμοποιούμε, να ξοδεύουμε τόσα πολλά κονδύλια, πριν πραγματοποιηθούν τέτοιε υποδομέ που έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον, γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια ανάλυση κόστου-οφελία. Είπαμε ότι θα την κάνουμε με διαφάνεια. Όταν θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα, και ότι θα αναλάβουμε τις σχετικές ευθύνες για τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν. Σε ό,τι αφορά τα άλλα προγράμματα, όλα βρίσκονται στη φάση υλοποίησης. Ε, ο αυτοκινητόδρομος στο Μπρένερο, η ΤΑΠ και οι επιταχύνσεις στις επενδύσεις και στα εργοτάξια, των εργοταξίων θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, με ταχύτητα σε όλα τα σχετικά έργα. Και με συγχωρείτε, Πρόεδρε, που θα καταχραστώ το χρόνο σας, αλλά δύο κουβέντες και για την εξωτερική πολιτική. Μας λέτε πολιτική απομόνωση. Η Ιταλία λέει είναι σε πολιτική απομόνωση. Για την Βενεζουέλα εμπόδισε τη διαδικασία και παρέμεινε απομονωμένη. Προσοχή εδώ, προσοχή. Πάνω απ' όλα, η Ιταλία σε καμία περίπτωση δεν είναι απομονωμένη συνεισέφερε τα μάλλα και αυτό είναι γεγονός, στην ε, έκδοση των ακινοθέντων από την Ήπατη εκπρόσωπο. Στις 26 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις, ε, δήλω, ε, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι και τη δική μου η τοποθέτηση ήταν η καθοριστική σημασία για να προκύψει αυτό το ανακοινοθέν. Πολλοί θέλουν να γράψουν την ιστορία πριν γίνει. Καλό θα ήταν εδώ να φανούμε συνετοί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση στην κρίση της Βενεζουέλας. Η Ιταλία ξέρει πολύ καλά τι κάνει και δεν είναι η μόνη. Είναι πολλές άλλες οι χώρες που έχουν ξεκάθαρες απόψεις. Ξέρουμε τι γίνεται και το θυμίζω για μας οι προεδρικές εκλογές του 2018 στη Βενεζουέλα δεν ήταν δημοκρατικές εκλογές, δεν τις αναγνωρίσαμε. Ναι, και επίσης ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζονται νέες προεδρικές εκλογές στη χώρα. Χρειάζεται να γίνουν με συνθήκες νομιμότητας, με διαφάνεια, να είναι αξιόπιστες βάσει των διεθνών προτύπων. Τις θέλουμε όσο δυνατόν νωρίτερα. Ε, γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που υποφέρουν και ήδη έχουμε προβλέψει από τα κονδύλια για καταπήγουσε ανθρωπιστικέ ανάγκε σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα να στείλουμε ποσά. Γνωρίζουμε ότι κανένα καθεστώ δεν μπορεί να δικαιολογεί την ύπαρξή του με τι βίε ενέργειε, με την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων με βία. Όμω, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε και να παρέμβουμε δεν μπορούμε να στέψουμε και να αναγνωρίσουμε κάποιον ο οποίος δεν προέκυψε ως αρχηγός ε, κράτους ή κυβέρνησης από ελεύθερες ανεξάρτητες εκλογές. Θέλουμε να δημιουργηθεί ομάδα επαφή, μια μορφή διαμεσολάβηση όπου να συμμετάσχουν όλοι. Υπάρχει ιστορική ευθύνη εδώ. Ιστορική ευθύνη να πούμε ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποιον σε το αξίωμα ε, ει βάρο κάποιου άλλου. Φανταστείτε στι μεγαλύτερε διεθνεί κρίσει από ιστορική ε, σκοπιά ε, τι εξέλιξη θα είχαν αν δεν είχαν όλοι βιαστεί να αναγνωρίσουν κάποιον ε, πρωταγωνιστή και σε είπα το αξίωμα ενώ υπήρχε ο αντίπαλός του ακόμα ε, στο προσκήνιο. Εδώ λοιπόν ριζοσπαστικοποιείται η αντιπαράθεση. Το να αναγνωρίσει κάποιος τον ένα σημαίνει ότι υποχρεώνει τους διεθνείς πρωταγωνιστές στο, στα διεθνή πράγματα να πάρουν το μέρος του άλλου. Θα γίνει χειρότερη κρίση σε σχέση με αυτές που σέρνονται ακόμα στις σελίδες της ιστορίας μας. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη συζήτηση με τη διαδικασία Catch the Eye. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το πολύ στις 19.45. 50 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Όσο περισσότερο μιλάτε εσείς, τόσο λιγότερο θα μιλάνε οι άλλοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, Υπουργέ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλήσατε για δημοκρατία. Εδώ πέρα βρίσκεστε ίσως στο πιο δημοκρατικό θεσμικό όργανο, γιατί είμαστε αμέσω έρετοι από τους ε, πολίτες. Σε αντίθεση με εσά ε, που διοριστήκατε. Εγώ είμαι περήφανη που είμαι Ιταλίδα, είμαι στο πλευρό της Ιταλίας, αλλά της Ιταλίας στην Ευρώπη. Και κοιτάξτε, ε, μας είπατε ότι υπάρχει ακριβώς ε, το θέμα θα είναι περίπατος ε, το θέμα αυτό του Made in Italy, η μεταρρύθμιση του Δουβλίνου κτλ. Ότι μας λέτε εργαστήκατε και έχετε κάνει συμμαχίε. συμμαχίε που δεν υπάρχουν στην Ιταλία, συμμαχίε που δεν υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μιλάτε για την Ευρώπη, μιλάτε για ενότητα και μετά μας λέτε ότι δεν θα κάνετε το τρένο, το ΤΑΒ. Δεν ξέρω αν ε, κάνω λάθος. Μετά μιλάτε για μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και ακούμε συνεχώς ότι τα πράγματα αυτά θα γίνουν προαιρετικά. Μα ε, τι αλληλεγγύη ε, μιλάμε μετά και τι αλληλεγγύη ζητάτε όταν θέλετε να είναι προαιρετικά. Είναι λοιπόν δικό σας το λάθος και καταλήγω το βίντεο σας με την καγκελάριο Μέρκελ είναι ντροπή γιατί εγώ αγαπάω την Ιταλία και δεν θέλω να κακολογεί ε, ο Πρωθυπουργός στην Ιταλική κυβέρνηση σε μια ομολογό του. Σας ευχαριστώ, Γκυγιόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε τη Κυβέρνηση, όταν δεν είμαι στο στραβού και τη Βρυξέλλε, ζω στη Λιόν. Είναι μια πόλη που έχει αρχαίου δεσμού με την Ιταλία. Είναι πολύ κοντά στο Πιεμόντε και βεβαίω το 16ο αιώνα ήταν πολλοί Λιονέζοι που μετανάστευσαν στην Ιταλία και αντιστρόφω πολλοί Ιταλοί μετανάστευσαν σε εμά. Και στο Τωρίνο, ε, τον αυτοκινητόδρομο που θέλουμε να φτιάξουμε το Ρήνο Λιόν, πώ γίνεται ακόμα να είναι στα χαρτιά. Δεν είναι απλώ για να συνδέσουμε δύο πόλει, είναι γιατί και το Καλέ από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει ένα δρόμο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το θέμα τη λεκάνη τη Μεσογείου και την διασύνδεση ε, μεγάλων πόλεων μεταξύ του. Μιλάμε λοιπόν για δεσμού. Ε, υπολογίζουν όλοι τα λεφτά, έχουν κάνει οι λογιστέ του απαραίτητου υπολογισμού και έχουν δει τι θα κοστίσει αυτό στο Ιταλικό κράτο. Σίγουρα σε πρώτη φάση τα έσοδα θα είναι λιγότερα από τα έξοδα και θα υπάρχουν οι φόροι του καυσίμων, λιγότερε οδικέ μεταφορέ, λιγότερα φορτηγά, λιγότερη ρήπανση. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξή. Δεν πιστεύετε ότι ο αδερφικό και παλιό δεσμό που ενώνει τι δύο χώρε μα δεν πρέπει να πάρει και πολιτική έκφραση, ε, ώστε να μην εμποδιστεί από ιδεολογικέ περιβαλλοντικές μέρημνε. Ευχαριστούμε κύριο κύριος Λούκερ. Κύριε Πρωθυπουργέ, σα ευχαριστώ για τι δηλώσει σα. Μίλησατε πολύ για αλληλεγγύη που ζητάει τώρα η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η συνεισφορά σα αυτή στο μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. ότι ζητάτε ε, αλληλεγγύη. Αλλά όταν μιλάμε για αλληλεγγύη πρέπει να μιλήσουμε και το γιατί καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση όπου αναγκάζει την Ιταλία να ζητήσει αλληλεγγύη. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από 20 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια, έχουμε ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ. Και εδώ και 15 χρόνια η Ιταλία δεν έχει καμία ανάπτυξη. Έχετε σκεφτεί μήπως υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δύο. Μήπως η Ιταλία θα έπρεπε να σκεφτεί αν κάνει αυτό το νόμισμα για τη χώρα θα μπορούσε, δεν ξέρω, η Ιταλία διαφορετικά να δημιουργήσει ένα έλλειμμα target 400 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μήπως οφείλεται εκεί στο ότι η Ιταλία συνεχώς παραβιάζει τους κανόνες ε, για το έλλειμμα. Κύριε Κόντε, όταν ζητάτε αλληλεγγύη πρέπει να τηρεί και τους κανόνες η Ιταλία. Στο σύστημα του ασύλου δεν το κάνετε. Πρώτα απ' όλα δεν τους καταγράφετε όλους και τώρα κλείνετε όλα τα λιμάνια και έχετε πάει στο άλλο άκρο. Λοιπόν, αν θέλει να είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Ιταλία, πρέπει να τηρεί του ευρωπαϊκού κανόνε. Αλλιώ δεν μπορεί να υπάρξει αλληλεγγύη. Σα ευχαριστώ. Τάραντ. Ονορεύει Μιράντα. Μιράντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ Κόντε, γιατί εμπόδισε η κυβέρνησή σας ένα σκάφος διάσωσης να ελιμενιστεί το 2018. Εγώ με τέσσερις ευρωβουλευτές του Κοινοβουλίου ε, επισκέφθηκα την Ιταλία και δεν πήραμε επίσημη απάντηση. Ο Υπουργό Μεταφορών σα είπε ότι πρόκειται για θέματα δημοσία τάξη και τέτοιου λόγου που εμπόδισαν τον ελιμενισμό. Ε, οι εκπρόσωποι τη Ιταλική κυβέρνηση ε, δεν μπορούσαν να μα εξηγήσουν γιατί έκτοτε μπλοκάρονται τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Γιατί μιλάτε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όταν δεν σέβεστε του κανόνε. Κανόνε αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, Σοκάρει το γεγονό ότι από στόματο ε, τη επίσημη κυβέρνηση, που θα μπορούσε να είναι πιο δημοκρατική, υπάρχουν διασυνδέσει με την ακροδεξιά, με φίλου του φασισμού, με φίλου όσων είναι αντίθετα με όσα προσβεύει η Ευρώπη. Ε, ο κύριο Μποργκέτσο. Στο νέο αρχηγό της κυβέρνησης Πρέπει να πω ότι προσφέρατε και πάλι αξιοπρέπεια σε μια χώρα που δεν ήταν συνηθισμένη σε αυτό. Ε, ένα λαό που, δεν είχε, συνηθί... που είχε συνηθίσει μάλλον να βλέπει ε, κολλημένου στον τοίχο του εκπροσώπου του όταν έρχονταν στην Ευρώπη. Καταφέρατε να πετύχετε πολλά ενώ υπήρχε η τάση ρήξη σε μια χώρα, σε μια χώρα καταφέρατε να, ε, να δείξετε ανάγλυφα την αλήθεια, την αλήθεια των γεγονότων, ότι η χώρα μας είναι μια μεγάλη χώρα όπου όλοι δουλεύουν σκληρά και ότι είναι σημαντικό να υπάρχει χρηματοδότηση, να στηριχθεί η οικονομία. Ζηλεύουν οι άλλες χώρες, ζηλοφθονία υπάρχει και πολλές φορές έχουν εκβιάσει ε, με, τις πολιτικές, με τα πολιτικά τους προσχήματα, προσπαθούν να περάσουν πολιτικούς στόχους και ευρωπαϊκούς, η οποία όμως είναι ουσιαστικά απόρρια χειραγώγησης. Σας ευχαριστώ λοιπόν που δείξατε τέτοια ε, σταθερότητα και στη συνεργασία με την άλλη συνιστόσα της κυβέρνησής σας που θέλει ε, να δείξει ότι η Ευρώπη είναι αρκετά απρόσεκτη, ότι το γεγονός ότι δεν καταφέρνει να εμποδίσει το εμπόριο ανθρώπων στην Μεσόγειο είναι ψεύδος και εξυπηρετεί άλλους σκοτεινούς σκοπούς. Η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, το εμπόριο αυτό εμποδίστηκε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την προσπάθεια που αναφέρατε να γίνει άνοιγμα προς τις αφρικανικές χώρες με τις οποίες πρέπει να υπάρξει διάλογος, να υπάρξουν συνθήκες αξιοπρέπειας και ισοτιμίας και εκεί και σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια ανοίγματο και συμμετοχή στο σύστημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας, στην υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο. Διότι μόνο σπήροντας έναν υγιή σπόρο, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πρόσφορο έδαφος, τότε θα προχωρήσουμε. Όχι αυτά που κάνανε οι παλιοί κυβερνώντες που πήγαιναν και άπλαναν τα πλοκάμια του στην Αφρική και κλέβαν από την Αφρική. Αυτό πρέπει να κάνει ένας αξιοπρεπής τίμιος λαός. Ευχαριστούμε κύριε Μπορκέτση, ο κύριος Βόιτ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε. Καταφέρατε να σταματήσετε αυτή την μαζική εισβολή μέσω της Μεσογείου. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Δεν είναι μυστικό ότι το λόμπι του ασύλου πλέον βγάζει λιγότερα λεφτά από ό,τι στο παρελθόν και το καταφέρατε εσείς. Και γι' αυτό κάνουν σαν να σας δικάζουν σήμερα. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι δικαστήριο. Τρίζουν οι παλιές ελίτ γιατί ξέρουν ότι σε τρεις μήνες δεν θα είναι πια η πλειοψηφία εδώ μέσα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, στη Γερμανία είδαμε ότι μπορούν και να σκοτώσουν οι μετανάστες κατά χιλιάδες. Σταματήστε τους φόνους και δώστε στα εκατομμύρια Ευρωπαίους που κοιτάνε σήμερα προς την Ιταλία και την Πολωνία την ελπίδα για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Χιμένες Πεσερίλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμερίζομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, αναχαιτήσουμε και να καταπολεμήσουμε το εμπόριο ανθρώπων στην Αφρική. Όμω δεν συμμερίζομαι την ουδετερότητα, τη στάση ουδετερότητα τη Ιταλία για το θέμα τη Βενεζουέλα. Διότι μπλοκάρατε την αναγνώριση του Γκουαϊντό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ την έχω την Ιταλία στην καρδιά μου. Έχω ε, παιδιά που είναι Ιταλοί στην εθνικότητα, στην Ιθαγένεια. Έχω ζήσει εκεί πάνω από 20 χρόνια και δεν καταλαβαίνω πως ένας Ιταλός δεν βλέπει την κατεπίγουσα ανάγκη ε, της ε, ε, Απομάκρυνση του κυρίου Μαντούρο που καταστέλει τα δικαιώματα των ε, κατοίκων τη Βενεζουέλας. Μιλήστε με τον κύριο Λόπε, μιλήστε με όλου του βασανισμένου, αυτού που έχουν βρεθεί στον τάφο, όλου αυτού του μετανάστε που βρίσκονται εκεί ε, και ζουν σε ένα φέρετρο στην ε, Κολομβία. Όπως είπε κάποιο, το μόνο απαραίτητο για να σταματήσει το κακό είναι να παραμένουμε αδρανείς. Είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος. Αναφέρομαι, ε, σας απευθύνομαι ως πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Στην ε, περιφέρεια μου παίρνουμε πολλά ε, εκατομμύρια ευρώ για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ιταλία. Για την παράκτεια και ορεινή όμως δράση μας δεν γίνεται τίποτα από την πλευρά της Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή θα σας θυμίσω την ανάκληση του πρέσβη ε, του πρέσβη μας μάλλον από τη χώρα σας και ότι πρέπει να υποστηριχθούν ξανά οι σχέσεις μας. Πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες διπλωματικές προσπάθειες που να δείχνουν ότι τα λόγια σας είναι πραγματικά υπέρ της Ευρώπης. Ε, στην ε, Γαλλία δείχνουν, φαίνεται ότι η πολιτική που χαράσουμε δεν μπορεί να συνδυαστεί με τη δική σας που απλώς μιλάει υπέρ της εθνικής κυριαρχίας της Ιταλίας και δεν έχει στόχο να είναι αποτελεσματική. Εάν θέλετε να υποστηριχθούν οι Ιταλοί φορολογούμε μόνο, θα αυτό θα είναι ει βάρο των Γάλλων πολιτών όμω και των Γάλλων ψηφοφόρων. Μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει προεκλογική εκστρατεία και ηθικέ ευθύνε. Με ένα φίλο σαν και εσά, τι να, τον κάνει, τι να κάνει κανεί του εχθρού. Η συμπεριφορά σα είναι άκομψη, αγενή, αφθάδη, ε, παράνομη και ε, συμμορήτικη. Θα πρέπει λοιπόν να ε, σα πω ότι δεν σα απευθύνω καμία αναγνώριση γιατί δεν σα αξίζει. Κυρία Τόγια. Ε, Πρωθυπουργέ, από τα λόγια των συναδέλφων εδώ ακούγεται πόση σεβασμός και εκτίμηση υπάρχει για την Ιταλία και πόση απογοήτευση και ανησυχία των φίλων μας για την Ιταλία. Πρέπει να τη δούμε πιο αντικειμενικά. Έχει αποδυναμωθεί, έχει απομονωθεί. Ε, υπάρχει διένεξη με τους συνεργάτες με τους οποίους θα πρέπει να χτίζουμε ένα κοινό μέλλον. Πώς μπορεί να είμαστε κατά της Ένωσης και της αλληλεγγύης. Εσείς τα είπατε, μόνο σας. Θα πρέπει λοιπόν με ευφυΐα και ε, ε ξυπνάδα να ε, ε, αρπάξουμε αυτέ τι ευκαιρίε. Και το λέω με απογοήτευση και όχι με χαρά, γιατί θέλω η Ιταλία, η χώρα μου, να είναι πρωταγωνίστρια στι μελλοντικέ εξελίξει. Και κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να ξεφύγουμε από τα πατηλά όνειρα και τι μεγάλες, ε, ε, ε, τα μεγάλα οράματα και τις χήμερες για το τι θα γίνει στη Μεσόγειο. Εδώ πρέπει να αλλάξει η στάση μας. Πού είναι η συνοχή για την οποία μιλάτε. Θα σας πω δύο πράγματα. Δεν λέω ότι τα καταφέραμε εμείς, γιατί η Ιταλία δεν φεύγει τώρα από την Ευρώπη. Αλλά να σα θυμίσω τα εξή και πείτε μου αν αυτή η εξοπιστία είναι ευρωπαϊκή, κύριε Πρωθυπουργέ. Για το κονδύλι για την Αφρική. Η πλειοψηφία σα ψήφισε κατά. Ε, για τα δισεκατομμύρια του προγράμματο Juncker. Τα δικά σα κόμματα που τώρα ε, κυβερνούν ε, ψήφισαν κατά. Για την απέτηση τη ενισχυμένη συνεργασία. Γιατί η Ιταλία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία των 9. Κατά. Για τι αρνητικέ συνέπειε του Brexit. Δεν ξέρετε ότι το μεγαλύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ιταλία είναι αυτό του Φάραντ. Μέσα από το δικό σα σα στο ε, διάβλο. Ε, κυρία Τόγια, κυρία Τόγια, παρακαλώ. Σα παρακαλώ λοιπόν να τρέψετε στην Ιταλία να ξαναγυρίσετε στη σωστή τροχιά. Ευχαριστούμε ο κύριο Ρανζέλ. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, προφανώς ε, με, το λόγο σας που ακούσαμε εδώ και με την τεράστιο σεβασμό που σας απευθύνουμε πρέπει να πω τα εξής. Ένα σημείο θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ θα πρέπει να θυμίσω τον Έλτο Μόρο και να θυμίσω ότι η τωρινή κυβέρνηση τη, ε, δεν θα πρέπει να θάψει τη μνήμη του Αλντομόρο και την φιλευρωπαϊκή του στάση. Δεν αρκεί όμως να τον αναφέρουμε σε σχέση με τη Μεσόγειο, πρέπει να τον αναφέρουμε και σε σχέση με την Ευρώπη. Ε, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι ω Πορτου... Πορτογάλο ευνηδιάζουμε από τη στάση τη Ιταλική κυβέρνηση στα θέματα τη Βενεζουέλα. Όχι απλώ γιατί θέτει ένα αμφιβόλο το όλο θέμα τη ευρωπαϊκή εξωτερική δράση, αλλά γιατί υπάρχει πορτογαλική κοινότητα στο Καράκα, στη Βενεζουέλα και υπάρχει και μεγάλη κοινότητα Ιταλών. Η Ιταλική κυβέρνηση δεν σκέφτεται του Ιταλού που ζουν και υποφέρουν λόγω του καθεστώτο του Μαδούρο, γιατί έχουν να υποστούν τα βασανιστήρια που του επιβάλλουν αυτή είναι η ερώτησή μου προ την Ιταλική κυβέρνηση. Ήδη θα έπρεπε να είχατε τοποθετηθεί. Δεν αρκεί να απαντήσετε τώρα. Έπρεπε να έχετε απαντήσει στην πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη. Μικρόφωνο. Έχω μία ερώτηση κύριε Πρωθυπουργέ. Πώς ε, βλέπετε ότι θα γίνει η κοινότητα, μια κοινότητα αλληλεγγύης ε, στα θέματα της ε, μετανάστευσης, πώς είναι δυνατόν να μας πηγαίνετε προς μια κατεύθυνση που, που επευλήθηκε στη Γερμανία με τους νόμους Χάρτς 4. Πώς είναι δυνατόν να σας επιβάλλουν τα πέντε αστέρια την ατζέντα τους στα κρίσιμα ζητήματα. Και είναι σοβαρά αυτά τα ερωτήματα, γιατί ακριβώς τη στιγμή που η Λέγκα αγκαλιάζει τις δυνάμεις της άκρας δεξιάς που θέλουν να πέσει η κυβέρνηση, μιλάτε ακριβώς για αλλαγή καθόλτος στην ε, Βενεζουέλα. Λοιπόν, σε τι βασίζεστε ως πρόβλεψη και ως ε, μελέτη ότι φέτος και τα επόμενα χρόνια θα είναι θαυμάσια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα μια απάντηση. Ο κύριος Σαλίνη. Πρόεδρε, καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα φανώ πραγματιστή. Ε, θα ήθελα να έχω χρόνο για να περιγράψω τι ε, κόπο έχει προκαλείται, ε, μάλλον με τι κόπο ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καταφέρουν να αποσπάσουν εκατομμύρια κονδύλια για τα έργα και τα προγράμματα που εκτελούνται στι διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε, μεταξύ των οποίων η δική μου. Θα χρειαζόμουν πολύ χρόνο για να αφηγηθώ πώ προσπαθήσαμε μέσα στο πέρασμα του χρόνου να δημιουργήσουμε σοβαρά προγράμματα που να συνδυάζουν τι απαιτήσει διασύνδεση τη χώρα μα τι απαιτήσει των επιχειρηματιών μα. Θα ήθελα να τα θυμίσω όλα αυτά και να αφηγηθώ κιόλα ε, σε τι ψυχική κατάσταση βρίσκονται όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ο ίδιο Υπουργό των Υποδομών και ότι ασχολείται περισσότερο με τις ε, χημικές ε, ε, με τα χημικά απόβλητα παρά με αυτές τις ε, περιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν ο, η κυβέρνησή σας να μας αποδείξει τις τεράστιες δυνατότητές της τις οποίες διαφημίζετε. Εγώ θα σας προκαλέσω στο εξή. Ε, πολλοί έχουν, προκαλέσει το, έχουν απευθύνει προκλήσεις σε κυβερνήσεις με, για πολιτικούς σκοπούς με αντικείμενο τους μισθούς. Εάν θέλετε λοιπόν να κάνετε μια αλλαγή στη χώρα, προβλέψτε ένα αντασφαλιστικό δάνειο ε, με σταθερό επιτόκιο και επιστρέψτε από τη δική σας την τσέπη για να δούμε πώς θα γεμίσουν τα ταμεία της χώρας μας. Ευχαριστούμε ο κύριος Βιώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρωθυπουργέ Κόντε, θα σας πω κάποια, κάποιους αριθμούς που είναι βαρετά ίσως. 2 ε, στα 6, 3 στα 4 για τον Σαλβίνη ε, ψηφοφορία λοιπόν. Ε, αποτελέσματα ψηφοφοριών ήταν αυτό και αυτές είναι οι απουσίες των Υπουργών της Ιταλίας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για νέους, μιλάμε για μηχανία, για μεταφορές, για μετανάστευση. Δεν είστε εκεί. Δεν είστε στι συνεδριάσει του Υπουργικού Συμβουλίου. Ζητήστε συγγνώμη από του Ιταλού. Ζητήστε συγγνώμη από του πολίτε τη Ιταλία και τη Ευρώπη. Δεν είναι αυτό η Ιταλία. Η Ιταλία χρειάζεται κυβέρνηση που να είναι παρούσα στην Ευρώπη. Να τη χρειαζόμαστε. Αυτέ τι δικαιολογίε που μα λέτε σήμερα, Πρόεδρε Κόντε, θέλουμε να ακούσουμε. Θέλουμε να είστε παρόντε πάνω απ' όλα. Και να κλείσουμε ένα παράθεμα. Ε, το είπατε κι εσεί, Πρόεδρε από το τραγούδι που κέρδισε το φεστιβάλ του Σαρέμο, του Μαμούτ, ε, ότι είναι δύσκολο κανείς να αλλάξει τον κόσμο αν δεν έχει καμία περηφάνεια. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η Ιταλία ε, δεν έχει πια τίποτα για το οποίο να είναι περήφανη Κοιτάξτε πώς είναι αδιαίθουσα. Παρακαλώ να χρησιμοποιείτε γλώσσα δέουσα και πρέπουσα για την Σύνοδο τη Ολομέλειας, ιδάλλως θα προβλέψω κυρώσεις για τους βουλευτές που χρησιμοποιούν ε, διατυπώσεις που δεν είναι κόσμιες και δεν αρμόζουν στο χώρο του Κοινοβουλίου. Δεν θα το ξαναπώ. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρωθυπουργέ της Ιταλίας, κύριε Κόντε, Μεσχέ Κόντε, Σενιόρε Κόντε, αν μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά. Can I start from the beginning, Mr. Chairman? Can I start from the beginning, Mr. Chairman? Κύριε Κόντε, είμαι σύμφωνος με αυτά που λέτε για την πορεία της Ευρώπης. Αλλά η Ευρώπη πρέπει να δείξει αλληλεγγύη. Και η αλληλεγγύη πρέπει να εκφραστεί και στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, στον τομέα της ασφάλειας. Και γνωρίζετε ότι η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα συνεχίζει να απειλεί την κύπρο παραβιάζει συνεχώς τον εναέριο χώρο της ελλάδος παραβιάζει τα χωρικά ύδατα της ελλάδος παραβιάζει την αόζ της κύπρου και θέλω μια δήλωση δική σας στήριξης της ελλάδος έναντι των απειλών της τουρκίας μια δήλωση δική σας που να στηρίζει την κύπρο να μπορεί να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους τη στιγμή μάλιστα που η ιταλική εταιρεία η eni θέλει και αυτή να αξιοποιήσει και να συνεργαστεί με την κύπρο για αξιοποίηση των φυσικών πόρων και απειλείται και η ιταλία και η ένι και η κύπρος από την τουρκία. θέλουμε μια δήλωση δική σας εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στήριξης της ελλάδας και της κύπρου και καταδίκης των απειλών του ερντογάν και της τουρκίας κύριε πρωθυπουργέ. το περιμένει ο ελληνικός λαός το περιμένουν επίσης οι φίλοι μας στην κύπρο. θέλουμε δήλωση συμπαράστασης. Καλώ Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να μπορείτε να με ακούτε. Ε, ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ, που ήρθατε. Ήταν έκπληξη. Θετική να σας ακούω. Και όπως λέμε στην Ίστρια, ε, θα πρέπει να μην ε, πουλάμε φύκια για μεταξωτέ κορδέλε, θέλουμε και γεγονότα. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε μια καλή συνεργασία και για την ιδιατρική. Με ενδιαφέρει να μου πείτε πώ βλέπετε τι σχέσει με τη Σλοβενία και την Κροατία και πώ βλέπετε να διαμορφώνετε το μέλλον για την συνεργασία με την Αδριατική. Είναι σημαντικό να μου πείτε πώ βλέπετε τη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τα Δυτικά Βαλκάνια. Και επίση με ενδιαφέρει αν η κυβέρνησή σα θέλει να περικόψει κονδύλια για τι Ιταλικέ μειονότητε, ε, για τη διγλωσία κύριε Υπουργέ Πρωθυπουργέ, ε, πρωθυπουργέ μάλλον, για την οποία εργάστηκα εγώ με συναδέλφου μου, ε, για την διγλωσία στην ε, Σλοβενία και την Κροατία. Χρειαζόμαστε χρηματοδόσει και από την Ιταλία, λέει ο μιλητή, στην Σλοβενία και την Κροατία. Θα μπορούσε να υπάρξει και ειδική σύνοδος που να ασχοληθεί με τα θέματα που αφορούν τους μετανάστες και τους ε, κατοίκους των άλλων χωρών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πενέσατε ε, και μιλήσατε για την σημασία τη ελεύθερη κυκλοφορία. Θα συμφωνήσω. Είμαστε η μεγαλύτερη γλωσσική γενιμονότητα που ζει στην Ιταλία κοντά στα σύνορα. Όμω η κυβέρνησή σα ε, έχει προβλέψει νόμο, το λεγόμενο Διατάγμα για την Ασφάλεια, που έχει να κάνει με πολλά άλλα, κυρίω με τη μετανάστευση και δεν θέλω να το σχολιάσω. Όμω βάσει αυτού του διατάγματο, εάν ένα φοιτητή ή κάποιο που θέλει να εργαστεί στο εξωτερικό πάει στο εξωτερικό, αγοράσει ένα αμάξι και θέλει να γυρίσει στην Ιταλία, το αμάξι αυτό θα το, το κατασχέσουν στα σύνορα και θα πληρώσει και 500 ε, ευρώ πρόστιμο. Μπορείτε να μου πείτε ένα τέτοιο μέτρο συνάδει με το μεγάλο ιδεώδες της ελεύθερης κυκλοφορίας που προσπιστήκατε. Ευχαριστούμε κύριο Σταραμπέλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να σας απευθυνθώ σήμερα, διότι ο κύριος Σαλβίνη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής σας που ήταν πριν από λίγο καιρό εδώ στο Κοινοβούλιο, μας είπε τις απόψεις του για τους πολίτες, αλλά μακριά από τις κάμερες. Ελεύθερα, λοιπόν. Θα Ήθελα να μου πείτε λοιπόν για αυτό τον τρόπο δράση ε, στην κυβέρνησή σα. Λίγα γίνονται και πολλά ε, ακούγονται ιδίω σε επίπεδο φιλιαρία. Επίση, πολύ εύκολα δακτυλοδεκτούνται οι ένοχοι για όσα σημαίνουν την Ιταλία. Πρόσφυγε, Αφρικανοί, ε, ομοφυλόφιλοι, Γάλλοι, η ίδια η Ευρώπη. Ε, κάποια στιγμή οι ένοχοι ήταν οι Εβραίοι και οι κομμουνιστέ, οι, οι Τσιγκάνοι, Αθήγανοι. Είναι τρόπο αυτό ε, να κάνει κανεί πολιτική. Δεν θυμίζει το φασισμό. Ε, αυτό κατέστρεψε την Ιταλία. Ε, ανάγκασε ε, εκατομμύρια Ιταλούς μετά τον πόλεμο να μεταναστεύσουν για να ζητήσουν το μέλλον του. Σα παρακαλώ, μην το λησμονείτε. Ο κύριος Τσίκου. Ε, Σα ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η χώρα, η χώρα μας περνάει μια φάση ύφεσης και δεν άκουσα κύριε Πρωθυπουργέ δυστυχώς να μιλήσετε για τη βιομηχανική πολιτική, την εμπορική πολιτική δεν άκουσα να μιλήσετε για τις επιχειρήσεις μας οι εμπορικές συμφωνίες ε, που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σημαίνουν ε, βεβαίω ε, εξαγωγές, εισαγωγές και ανάπτυξη θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί η φορολογία για να μπορέσουν να δώσουν δουλειέ οι επιχειρήσεις μας και να, να σταματήσουμε τις επιδοτήσεις που δεν χρησιμεύουν ε, σε τίποτα παρά να παριστάνουμε ότι καταπολεμούμε την φτώχεια και την ανισότητα. Σας παρακαλώ λοιπόν να μου δώσετε μία απάντηση. Σας ευχαριστώ Μπρέσο. Κύριε Πρωθυπουργέ, όπως ε, ήδη κάποιοι συνάδελφοι είπαν και όχι μόνο οι Ιταλοί, εμείς εδώ εργαζόμαστε σε έργα που στόχο έχουν να βοηθήσουν την Ιταλία και την Ευρώπη. Και η γραμμή αυτή, η μεταφορική ε, της Μεσογείου, γιατί δεν είναι μόνο από το Τωρίνο στην Λιόν, είναι αυτή ακριβώς η οποία θα αποκαταστήσει την ισορροπία του συστήματος μεταφορών προς Νότον και όταν ολοκληρωθεί θα συνδέσει τα λιμάνια της Μεσογείου και θα επιτρέψει να αναπτυχθούν. Και το είπατε επίσης ε, ότι η κυβέρνησή σας ε, έχει κάνει μία ανάλυση κόστος ωφέλους η οποία όμως δεν λαμβάνει υπόψη το χρονικό πλαίσιο σε βάθος 50 ετών ε, για την απόσβεση Κύριε ε, Πρωθυπουργέ, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να σκέφτεστε μόνο και σαν Ευρωπαίος και όχι μόνο να σκέφτεστε τα μικρά εσωτερικά ιταλικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ, ε, εγώ θα σας πω ότι είμαι από την Σουηδία, μεν εκλεγμένη, αλλά είμαι περήφανη που είμαι Ιταλίδα. Αλλά ε, τώρα πια είμαι όλο ένα λιγότερο περήφανη για την Ιταλία μου. Την Ιταλία που εργάζεται, που έχει τεράστια καραδιά, ε, που δεν γυρνάει τις πλάτες όταν τα παιδιά βρίσκονται να κολυμπάνε στη θάλασσα, που κλείνει τα λιμάνια της, που γνωρίζει ότι το κοινό μας μέλλον είναι η Ευρώπη. Εδώ και ένα χρόνο η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος, την αξιοπιστία της σε όλα τα μέτωπα. Ανησυχεί η ε, ε, κακοδιαχείριση της οικονομίας που έχει φέρει σε ύφεση την Ιταλία. Οι νέοι, κύριε Πρωθυπουργέ, οι νέοι ζητούν δουλειά, δεν ζητούν ελεημοσύνη. Θέλουν αξιοπρέπεια και όχι κουβέντε προπαγάνδα. Θέλουν συγκεκριμένε απαντήσει. Τι θα δώσετε συγκεκριμένε απαντήσει μα ακούτε, στις, ε, στους ε, στην ελάφρυνση του χρέου που οδηγεί στη φτώχεια οικογένειε και επιχειρήσει. Με ακούτε. Α, ωραία, ευχαριστώ. Ε, και ανησυχεί ακόμα περισσότερο ε, ο εκτροχιασμός προς την εθνική κυριαρχία και τον εθνικισμό της κυβέρνησής σας. Δεν είναι το πρόβλημα η συνεργασία της Ιταλίας με άλλες χώρες. Η Ιταλία είναι μια χώρα σε θέση να χτίζει γέφυρες, όχι να ανοίγει χαντάκια και ε, να προκαλεί ρήξεις. Χρειάζεται αλληλεγγύη αλλά με διάλογο, όχι με προσβολές πα, πα, ε, φτάνει αυτή, αυτό το παράδοξο που λέει ότι οι γειτονέ μα είναι οι πρώτοι μα εχθροί. Δεν θα προχωρήσουμε αν δεν δημιουργούνται ε, συμμαχίε. Ε, δεν θα δημιουργήσουμε σωστά. Μα μας ακούν ο Γκάσπαρη και ο Σπινέλη και μα βλέπουν. Αλλάξτε πορεία, κύριε Κόντε. Σόλτε. Κύριε Σόλτες. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μιλήσω για μια αλληλέγγυα Ευρώπη, μια Ευρώπη της συμφιλίωσης, μια Ευρώπη ενωμένη. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και εσείς ο ίδιος μιλάτε με λόγια που δείχνουν το μίσος σαν τα θύματα να μην ήταν αρκετά στο παρελθόν. Αρνείστε με κάποιο τρόπο την ιστορία. Τα θύματα αυτά έδωσαν τη ζωή τους έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά συμπεριλαμβανομένου και το σύνορο μεταξύ Σλοβενίας και Ιταλίας και πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να παραιτηθείτε μετά από αυτά στη σχόλια. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. κυρία Σλάιν δεν μπορώ να του ικανοποιήσω όλου. Είναι 50 οι βουλευτέ. Έδωσα και παραπάνω χρόνο. Ο καθένα θέλει να μιλήσει. Κύριε Κόντε, παρακαλώ. Απαντήστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ορισμένες παρεμβάσεις έθιξαν θέματα πολιτικού χαρακτήρα. Η πολιτική συζήτηση σκοπό έχει να εξυπηρετεί την ε, δημοκρατική λειτουργία. Ε, ακόμα και αν είναι εντονή, ακόμα και αν κάποιε φορέ είναι δυσάρεστε οι αντιπαραθέσει. Κάποιε παρεμβάσει δεν θα πρέπει καν να σχολιαστούν. Διότι προφανώ νομίζουν ότι θα προσβάλλουν όχι μόνο τον ίδιο τον ομιλόντα, αλλά τον ολόκληρο, το λαό που εκπροσωπεί. Που εγώ εκπροσωπώ. Ορισμένοι είχαν το θράσος, και το λέω με απόλυτη επίγνωση, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κάποιοι είπαν και ως επικεφαλής ομάδας, εκπροσωπώντας ολόκληρη πολιτική ομάδα, ότι είμαστε παλιάτσι που εκπροσωπούμε τον Ιταλικό λαό. Εγώ δεν είμαι μαριονέτα, δεν είμαι μαριονέτα ούτε αισθάνομαι έτσι. Είμαι υπερήφανο που εκπροσωπώ έναν ολόκληρο λαό. Είμαι υπερήφανο και καμαρώνω που μπορώ να ερμηνεύσω τη βούληση για αλλαγή των Ιταλών και, των... και ολόκληρου του λαού. Είμαι υπερήφανο που μπορώ να συγκεφαλαιώσω την πολιτική γραμμή μιας κυβέρνησης που δεν είναι μαριονέτα, γιατί δεν ακολουθεί λογικές των λόμπι, ούτε επιχειρηματικών κύκλων. Ίσως μαριονέτες είναι αυτοί που ασχολούνται με τα λόμπι, τις επιχειρηματικούς ομίλους και τις τραπεζικές ομάδες μου είπατε ορισμένοι και νομίζω και εδώ ε, ξεφεύγουμε από την έντιμη και έστω και ε, δύσκολη πολιτική συζήτηση ότι υπάρχει ε, και μια κουβέντα που έγινε μεταξύ μου και της καγκελαρίου Μέρκελ Όποιος ε, τα είπε αυτά μπορεί να ντρέπεται δημοσίως για δικό μου λογαριασμό αν ίσχυαν αυτά τα λόγια. Είπε ότι εκπρόσωπος ενός ε, έχει υψηλά ρεκόρ ε, ως προς την ε, ε, εκτίμηση που του τρέφει το κοινό. Ίσως άλλοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ντρέπονται μεταφέροντας αυτά τα λόγια. Επίσης και εδώ φτάνουμε στο τρίτο σημείο που κατά την άποψή μα ε, ξεφεύγει από την έντιμη πολιτική συζήτηση, ακόμη και αν αυτή ήταν ε, έντονη, ότι οι υπουργοί μου υπόθηκε μάλλον ότι οι υπουργοί μου δεν συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Υπουργικά Συμβούλια. Η κυβέρνησή μου δεν παρίσταται στη συνόδους των, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν θα σα θυμίσω τι γίνεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Απλώ να θυμίσω ότι η κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπηθεί και από υφυπουργό, από κάποιον άλλο εκπρόσωπο και ότι ανέκαθεν παριστάμεθα σε όλε τι συνόδου και σε όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια και συμβούλια υπουργών. Το θυμίζω και το τονίζω για να είμαι ακόμη πιο άμεσο και ότι εσείς που εκφράζετε ένα κόμμα το οποίο στο παρελθόν δεν ε, συμμετείχε επαρκώς στην περίπτωση της αίμα και ακόμα πληρώνουμε τις συνέπειες. Ε, κατά τα άλλα, Πρόεδρε, θα έρθω τώρα στις ερωτήσεις. Vengo και τώρα έρχομαι. Κύριε Ντάντε, σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε λίγο διαφορετική γλώσσα. Ας προσπαθήσουμε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε δύο λεφτά. Παρακαλώ. Πρωθυπουργέ, με συγχωρείτε. Παρακαλώ όλες και όλους μην χρησιμοποιείτε προσβλητικέ εκφράσει. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, μπορείτε να εκθέσετε οποιαδήποτε πολιτική θέση σα αρέσει, αλλά μην προσβάλλετε του άλλου. Και άλλοι εκπροσωπούν ε, ε, το λαό και είναι νομίμω εκλεγμένοι. Μην προσβάλλετε τον Πρωθυπουργό τη Ιταλική Δημοκρατία, ο οποίο έχει προσκληθεί από εμά εδώ. Δεν έχει έρθει ε, με το ζόρι. Τον καλέσαμε. Σας παρακαλώ λοιπόν κόσμια γλώσσα απευθύνομαι κυρίω στου συμπατριώτε μου, του Ιταλού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ λοιπόν θα έρθω και στα πολιτικά ζητήματα που τέθηκαν, που είναι επίση πολύ ενδιαφέροντα να απαντήσω σε συγκεκριμένο αίτημα. Μου ρωτήθηκε να πω για την στήριξη προ την Ελλάδα και την Κύπρο. Να θυμίσω στι 29 Ιανουαρίου ήμουν στην Λευκοσία, όπου μαζί με άλλε 7 χώρε τη Νοτιού Ευρώπη ε, συζητήσαμε και δώσαμε και μια τελική συνέντευξη τύπου κοινή και είπαμε, τοποθετηθήκαμε συγκεκριμένα. Οπότε υποστήριξη προ την Κύπρο έχει ήδη δοθεί. Σε ό,τι αφορά τα άλλα ερωτήματα, ε, υπόθηκαν πράγματα πραγματικά που προκαλούν ντροπή για την Ιταλία. Ότι αφήνουμε να πεθαίνουν παιδιά στη θάλασσα. Αυτά είναι πραγματικά σοβαρά, είναι ε, απίστευτα αυτά που λέγονται. Το είπα και προηγουμένως έχουμε καθήκον να ενημερωνόμαστε όταν μιλάμε εδώ από αυτά τα έδρανα. Είπα προηγουμένω ότι ανέκαθεν ίσα ίσα που παρενέβημε... για να φροντίσουμε ότι ε, εξασφαλίζουμε την ακαιρεότητα των πιο ευάλωτων, ακόμα και σε δύσκολε και πολύ προβεβλημένε υποθέσει διάσωση. Κοιτάξαμε πρώτα την ασφάλεια γυναικών και παιδιών, του μεταφέραμε. Του ε, αποβιβάσαμε από τα σκάφη, τους του. Ε, εδώ λοιπόν την αλληλεγγύη τη θεωρούμε κάτι που εκφράζεται στην πράξη. Στην Ευρώπη θα πρέπει να περάσετε από τα λόγια στα, στις, στη δράση. Ε, Όσοι χώρα έχουμε κάνει πολλά. Γαλλία, για το κεφάλαιο Γαλλία. Ε, το είπα επανειλημμένως η Ιταλία είναι υπερήφανη για τον παλιό της δεσμό, οικονομικό και πολιτιστικό κυρίως με τη Γαλλία. Ξεκινά με τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Ποιος το αμφισβητεί. Μιλάτε για διαφωνία, μιλάτε για αντιπαράθεση, για μια συγκεκριμένη υπόθεση και λέτε ότι πάει στην ουσία. Μιλάμε για δύο συστήματα που λειτουργούν παράλληλα και συνδυάζονται, ε, αλληλοδιεκτρέφονται στον, ε, αλληλοτροφοδοτούνται μάλλον στο πολιτιστικό επίπεδο και το οικονομικό. Επίσης, συζήτησα με κάποιους εκπροσώπους του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων Βεβαίως αυτό έγινε στα πλαίσια του ιδιότητα ενός ηγέτη πολιτικής ομάδας. Πρέπει να υπάρχει πολιτική συζήτηση. Πρέπει οι επιλογές να μπορούν να τεκμηριωθούν, ε, οπότε εφόσον τεκμηριώνονται είναι και νόμιμο, νόμιμες και θεμητές. Για τη Βενεζουέλα υπόθηκε κάτι που είναι κατάφορα ψεύδος. Ε, η Ιταλία υποστηρίζει το Μαδούρο και η Ιταλία δεν ζητά προεδρικέ εκλογέ. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. εδώ δεν υπάρχει ότι δεν βιαζόμαστε. Οι δηλώσει μου είναι όλε το αντίθετο, λένε. Το καθεστώ του Μαδούρο σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται από την Ιταλία. σα ίσα διακηρύξαμε ε, και αποφανθήκαμε ότι οι προεδρικέ εκλογέ δεν ήταν νόμιμε. Το Ευρωκοινοβούλιο τι αναγνώρισε. Δεν αποστήλαμε τίποτα ε, ω ε, αναγνώριση. Δεν θεωρούμε ότι ο πρόεδρο Μαδούρο έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Ζητάμε όμω το δυνατόν νωρίτερα προεδρικέ εκλογέ. Ελεύθερε. Και το έχουμε πει με κάθε τρόπο εκλογέ ω το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί ο πληθυσμό τη χώρα υποφέρει. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό θα ε, επιτευχθεί εάν ε, υπάρξουν ε, τέτοιε ρήξει στη χώρα και αναγνωριστεί, το είπα, το αξίωμα πρόεδρο κάποιο που δεν έχει κερδίσει νόμιμα εκλογέ. Πρέπει γρήγορα να πάμε σε ταχεία επίλυση του θέματο με δημοκρατικό τρόπο. Επίση, και νομίζω τέθηκε το θέμα της οικονομίας ρωτήθηκε γιατί η Ιταλία δεν δίνει σημασία και στην ευρωπαϊκή διάσταση της βιομηχανικής πολιτικής. Έχουμε αναγνωρίσει τη σημασία του προγράμματος Juncker, το είπα εγώ ίδιος. Ανέκαθεν υποστηρίζαμε την σημασία και την αξία μιας βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρώπη, από την Ευρώπη. Ε, μάλιστα, έχουμε υπογραμμίσει την σημασία ενό προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Ε, προπολογισμού που θα έχει και μια λειτουργία σταθεροποίησης και για να παραμείνουμε στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής και της κοινωνικής πολιτικής, η χώρα μας, κοιτάξτε, είπατε, δεν αναπτύσσεστε. Τι θα πει αναπτυσσόμαστε. Θα πρέπει να βασιστούμε σε πολιτικούς υπολογισμού του παρελθόντος. Μήπως είναι ακόμα λίγο νωρί. Μήπω είναι ακόμα λίγο νωρί για να αξιολογήσουμε ο οικονομικό ελιγμό που κάνουμε τώρα, η αλλαγή πορείας που ακόμα πραγματοποιείται, θα δώσει καρπούς. Εγώ έχω αναπτύξει ένα σκεπτικό ότι η οικονομική ανάπτυξη θα γίνει στο δεύτερο εξάμεινο, θα ξαφνιέται στο δεύτερο εξάμεινο το 2019, διότι ακριβώς και πολύ απλά η οικονομική μας πολιτική, τα μέτρα μας δεν μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως αυτούς τους πρώτους μήνες του έτους. Ε, να έχετε υπόψη ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά το σύστημα παραγωγής. Πώς θα μπορούσαμε να μην ασχολούμαστε με το πρόγραμμα επενδύσεων το είπα και προηγουμένως. Και κάποιοι είπαν κάτι εντελώ λανθασμένο. Βεβαίω και εργαζόμαστε από αυτού. Και χθε μόλι, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, εγώ ο ίδιο βρισκόμουν στην περιοχή τη Νότια Ιταλία, την περιφέρεια αυτή, όπου είναι μεγαλύτερη οικονομική ύφεση σε σχέση με αλλού, και για σκοπού κοινωνική ανάπτυξη υπέγραψα τρει ε, συμβάσεις στο Μολύζα, τη Σαρδινία και την Παζιλικάτα για σκοπούς κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό έχει πραγματιστικό σκοπό. Θέλουμε να στηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη με όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Ακόμη και το εισόδημα, το ελάχιστο εισόδημα για τους πολίτες, για τους φτωχότερους πολίτες. Θα μπορούσε να είναι σοσιαλιστικό τέχνασμα. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Όλοι το συζητάνε αυτό το μέτρο γιατί έχει καταλητικό χαρακτήρα για τις δημόσιες συζητήσεις. Εδώ όμω είναι υπαρξιακό το θέμα διότι είναι και θέμα προπολογισμού και κυρίως το συλλάβαμε στο επίπεδο ενός συμφώνου εργασίας, κοινωνικής συμπερίληψης, για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε στο χώρο της, αγο... της εργασίας και της παραγωγής 5 εκατομμύρια φτωχούς. 5 εκατομμύρια φτωχούς ε, στους οποίους απευθύνεται απευθείας αυτό το μέτρο είναι τελώ εκτό συστήματο, οποιοδήποτε κοινωνικού παραγωγικού μηχανισμού, ε, εκτό του χώρου τη εργασία. Χωρί το άρθρο 3, στο δεύτερο εδάφιο του υπέροχου συντάγματό μα, του συντάγματο τη Ιταλία, δεν θα έχουν καμία ε, ηλική, καμία χειροπιαστή πραγματικότητα να συμμετέχουν στην ε, δημοκρατική, κοινωνική και πολιτική διαδικασία και το γίγνεσθε τη χώρα μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ εγώ κύριε Πρωθυπουργέ, εκπρόσωπε του, της Ιταλικής κυβέρνησης, της ε, Δημοκρατίας της Ιταλίας. Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας και τις απαντήσεις σας. Με συγχωρείτε κάποιες φορές το ύφος που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν κατάλληλο, αλλά στην Ολομέλεια πάντοτε είναι έντονες οι συζητήσεις, γεμάτες πάθη, όταν υπάρχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα τα οποία συζητούμε. Πάνω από όλα σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ένωσής μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ πολύ αποχωρήστε ήσυχα όσοι αποχωρείτε. Σε σχέση με τις συστάσεις για απόφαση από την Επιτροπή Σύντερ και ΕΚΟΝ, ε, για να μην διατυπωθούν αντιρρήσεις σε πράξη κατά εξιοδότηση. Ε, είδαμε ότι δεν υπάρχει καμία αντιρρήση μέσα στις 24 ώρες που είχαμε δώσει ως προθεσμία, οπότε εγκρίνονται. ε, άρθρο 105, παράγραφος 6 λοιπόν του κανονισμού μας που λέει ότι πλέον στάσεις αυτές μπορούν να υιοθετηθούν επισήμως και θα δημοσιευθούν αύριο την Τετάρτη 13 ε, Φεβρουαρίου. Η συζήτηση ήταν φορτισμένη προηγουμένως, τώρα ας ηρεμήσουμε και ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέσιας διάταξης που είναι η κοινή συζήτηση Συμφωνία Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Σιγκαπούρη. Η συζήτηση θα γίνει επί τη βάση της έκθεσης του David Μάρτιν για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης. Επιπλέον έχουμε ένα ψήφισμα και μια σύσταση που αφορά την προστασία των επενδύσεων μεταξύ των δύο. Και άλλη μια έκθεση του κυρίου Μάρτιν και άλλο ένα ψήφισμα και μια σύσταση του κυρίου Ιστούρης. και άλλη μια έκθεση του Αντώνιο Λόπεση Τούρι Βάιτ ω ψήφισμα για την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Σιγκαπούρη. Ξεκινάμε τι συζητήσει. Καλώ ήρθατε κυρία Επίτροπε. Πρώτος ομιλητής θα είναι ο εισηγητή, ο κύριος Ντέβιτ ε, Μάρτιν. ναι,